darf sie bitten platz zu nehmen. η συνεδρία, η διάσκεψη των Προέδρων που σήμερα είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη ξεκινάει τώρα και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τίμερμαν, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το Κοινοβούλιο προετοιμάζει την ε, ψηφοφορία για τη νέα Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 115 και το παράρτημα 16 του κανονισμού. Προς αυτό έχουμε τα, τους προτινόμενους ε, υποψήφιους ε, επιτρόπους, ε, τους οποίους εξετάσαμε σε σχέση με τις ικανότητές τους και την ανεξαρτησία της σκέψης τους. Επίσης, οι γνώσεις τους για τον χαρτοφυλάκιο τους και οι δυνατότητες επικοινωνίας και αυτές πρέπει να αξιολογηθούν. Και προς αυτό θα εξυπηρετήσει η σημερινή ακρόαση, η οποία είναι και η τελευταία πριν από την αξιολόγηση που θα λάβει χώρα από τους Προέδρους των Επιτροπών. Ο κύριος Τίμεμανς θα προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση κατά το μέγιστο 15 λεπτών. Κατόπιν ε, θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Τίμερμανς, συνολικά 45 ερωτήσεις που θα υποβάλλετε εσείς αγαπητοί συνάδελφοι. Και για κάθε ερώτηση προβλέπετε κατά το μέγιστο ένα λεπτό. Ο κύριος ε, Τίμερμανς ε, για να απαντήσει θα έχει δύο λεπτά για κάθε ερώτηση. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα και ως προς τις ερωτήσεις παρακαλώ να εστιάζεστε σε σημαντικά θέματα. Αυτή λοιπόν η ακρόση μεταδίδεται ζωντανά ε, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άλλη μια τεχνική φύσεως παρατήρηση. Κυρίε και κύριοι, με γνωρίζετε, ξέρω ότι είμαι ένας πολύ φιλικός ε, και προσινής άνθρωπος, καλός άνθρωπος θα έλεγα, εκτός όταν πρόκειται για την υπέρβαση του χρόνου μιλίας. Και αυτό ως προς αυτό σήμερα θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρός γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί ο κύριος Τίμερσμαν να έχει χρόνο για να απαντήσει. Που σημαίνει ότι μετά από 15 δευτερόλεπτα θα αρχίσουν ε, να ανάβουν τα φωτάκια και μετά από 60 δευτερόλεπτα θα σας ε, παίρνω το λόγο. Λυπάμαι που ε, πρέπει να σας το πω ευθύ εξ αρχής, αλλά πραγματικά το εννοώ. Κύριε Τίμερμαν, εσείς έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν λοιπόν να τηρήσετε και εσείς ε, το χρόνο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσείς μπροστά σας ε, θα βλέπετε αυτά τα δύο κόκκινα στεράκια που τα αναποσβήνουν και θα δείχνουν ότι τελειώνει ο χρόνος σας. Ε, έχετε άλλες ερωτήσεις παρακαλώ, παρακαλώ επί της διαδικασίας. Όχι από